θα ήταν ε, εν τέλει καλό για, την Ευρωπαϊ... για το ε, Ηνωμένο Βασίλειο και δεν θέλουμε να είμαστε μέλος αυτού του πειράματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα τον λόγο έχει ο κύριος Μάρτιν Έρενχάουζερ. Κύριε Φάραντς,